Συνεχίζουμε την συνεδρίασή μας. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη Συμφωνία Προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Θα ξεκινήσουμε με τον ε, Υπουργό, τον κύριο Λοπές Καρίγκο. Έχετε το λόγο εξ του Συμβουλίου, κύριε Υπουργέ.